δηλώσει του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τις διατλαντικές ροές δεδομένων. Θα δώσω το λόγο και πάλι στον Υπουργό Κούντερς. Uh, Mr. President, yeah. uh, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε, η Προεδρία αποδίδει μεγάλη σημασία σε, μια ελεύθερη, σε ένα ελεύθερο, ανοιχτό και ασφαλές ίντερνετ. Και αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για μένα. Στην ψηφιακή εποχή είναι πολύ γνωστό ότι τα προσωπικά στοιχεία είναι μεγάλης αξίας λόγω των πληροφοριών που περιέχουν διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να προσωποποιήσουν ε, τις προσφορές τους προς καταναλωτές ε, και στις ε, αρχές επιβολής του νόμου να ανοιχνεύσουν τους εγκληματίες, καθώς και προσφέρουν διάφορες εμπορικές ευκαιρίες. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να προστατευτούν ώστε να προστατευτεί η ιδιωτική μας ζωή. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στις ροές δεδομένων, εμπιστοσύνη που βασίζεται σε ένα σωστό πλαίσιο προστασίας. Από μεταφορές ε, προσωπικών δεδομένων εκτός της Ένωσης, η διατλαντική ροή είναι η πιο σημαντική ε, με μεγάλη διαφορά. Είτε πρόκειται για εμπορικούς είτε για ε, αστυνομικού λόγους. Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης και των πολιτών της η ασπίδα Ένωσης και είπα να εξασφαλίζει αυτήν την εμπιστοσύνη και προστασία, ιδιαίτερα μετά την απόφαση του 10 τον περασμένο Οκτώβριο. Εξασφαλίζεται έτσι η κάλυψη για αυτό το τομέα που είναι τόσο ζωτική σημασία για την διατλατική οικονομία και αθώ και για τι μικρομεσαίες ευρωπαϊκέ εταιρείε που εξαρτώνται από αυτή την ε, απόφαση καταλληλότητα ώστε να εξασφαλίσουν την ασφαλή μεταφορά δεδομένων προ τη ΣΥΠΑ. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη πλήρω την απόφαση του δικαστηρίου για το καθεστώ ασφαλού λιμένα. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ένα επίπεδο προστασία δεδομένων που θα σέβεται τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τι συνθήκε καθώ και τα πρότυπα που ορίζονται από την πρόσφατη νομολογία. Οι ισχυρέ δικλείδε ασφαλεία αποτελούν το κλειδί για την αποκατάσταση τη εμπιστοσύνη του κοινού όσον αφορά τι διατλαντικέ ροέ δεδομένων. Το Συμβουλίο, το, εμείς, το Συμβούλιο εμπιστευόμαστε την Κομισιόν Κομισιόν ώστε να εξασφαλίσει τα ανώτερα δυνατά ε, στάνταρ ασφάλειας ε, εφαρμόζοντας ε, τον περιορισμό των, της, του στόχου χρήσης ή την αντίρρηση κατά της επεξεργασίας καθώς και ένα αποτελεσματικό σύστημα εποπτείας, επιβολής και δυνατότητας αποζημίωσης. Επιπλέον θέλουμε να παροτρύνουμε την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους ομολόγους της ΣΥΠΑ ώστε να βελτιώσει βελτιώσει κάποιε λεπτομέρειε τη ασπίδα και να εξασφαλίσει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Πιστεύω ότι η συλλογή από πλευρά τον είπα, θα μπορεί να είναι αποδεκτή μόνο υπό συγκεκριμένου όρου. Στο ίδιο πνεύμα, καλωσορίζω την ε, δημιουργία ενό διαμεσολαβητή, έναν επιπλέον μηχανισμό για το χειρισμό των ε, παραπώνων των πολιτών. Για την διατλαντική μεταφορά προσωπικών στοιχείων για εμπορικού σκοπού, το Συμβούλιο θεωρεί πω η Επιτροπή θα οφείλει να ε, υιοθετήσει την απόφαση περί καταλληλότητα σε αυτό το διατλαντικό πλαίσιο τάχιστα, ενώ εξασφαλίζει τα δικαιώματα Προστασία των δεδομένων των πολιτών. Εργαζόμαστε σε μια συμφωνία ώστε να, μάλλον, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ένωση και στη ΣΥΠΑ. Επίσης συνεχίζονται διαπραγματεύσεις ώστε οι Κομισιόν και οι εθνικές διοικήσεις να οδηγήσουν σε, ένα σε μια θετική έκβαση ε, δρομολογώντας ε, ε, την έναρξη ισχύω μια τέτοια συμφωνία. Το Συμβούλιο στοχεύει στο να υιοθετήσει απόφαση για να υπογράψει μια συμφωνία γενική, ε, ώστε να μπορέσει να υπογραφεί στην Υπουργική του Άμστερνταμ ένα σύμφωνο και θα ζητήσουμε μετά και την συγκατάθεση του Ευρωκοινοβουλίου για να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία δεν, δεν παρέχει βάση για την ε, μεταφορά των προσωπικών δεδομένων οργάνων στη διατλαντικά. Απλά θα θεσπίσει κοινέ προδιαγραφέ προστασία των στοιχείων. Ε, αυτό είναι καλά νέα από την ευρωπαϊκή προοπτική, γιατί οι ΙΠΑ δεσμεύονται να σεβαστούν υψηλότερε προδιαγραφέ από το παρελθόν όταν λαμβάνει προσωπικά στοιχεία από την Ευρώπη. Και αυτό είναι απαραίτητο. Έτσι, η συμφωνία θα συμβάλλει στην αποκατάσταση τη εμπιστοσύνη στι ροέ τη Διατλαντική για την, ε, τον στόχο τη καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων, προσθέτοντα ένα επιπλέον ε, επίπεδο προστασία των δεδομένων για την Ένωση και τη ΣΥΠΑ. Το Συμβούλιο θεωρεί πως η συμφωνία αυτή αποτελεί βελτίωση σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά την δικαστική αποκατάσταση ε, γιατί για πρώτη φορά οι ΗΠΑ δέχονται να επεκτείνουν αυτά τα δικαιώματα στους Ευρωπαίους πολίτες. Δηλαδή ένας Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να χαίρει ίσης μεταχείρισης και να έχει τα ίδια δικαιώματα δικαστικής αποκατάστασης όπως και ένας ε, Αμερικανός πολίτης. Ε, είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να συμφωνήσει μαζί μας αυτήν την αξιολόγηση. Εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλή ασφαλής μεταφορά προσωπικών στοιχείων προς τη ΣΥΠΑ. Εξασφαλίζουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, των πολιτών μας γίνονται σεβαστά στο ποινικό αλλά και στο ε, δίκαιο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία σε διατλαντικές ποινικέ έρευνε, Συλλέγονται τα στοιχεία ε, ε, και αν κάποιο πολίτη, Ευρωπαίου πολίτη το όνομα καταλήξει σε κάποια μαύρη λίστα θα μπορεί να ζητήσει αδίκως, θα δεν μπορεί να ζητήσει δικαστική αποκατάσταση. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα ότι δηλαδή θα υπάρχει ένα βελτιωμένο σύστημα εποπτείας και επιβολής που θα αυξήσει την αξιοπιστία του συστήματος στον τομέα της επιβολής του νόμου. Θα έχουμε πολύ αυστηρές προδιαγραφές ώστε να προβλέπεται και διόρθωση αποκατάστασης για όλα τα μέσα που καλύπτονται από την ευρύτερη συμφωνία. Ελπίζουμε πως η Κομισιόν γρήγορα θα λάβει μια απόφαση όσον αφορά την ασπίδα, θα σεβαστεί τι εκτιμένο Επίσης, είμαστε πεπισμένοι ότι η συμφωνία ε, ομπρέλα είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση, καθώς εισάγει νομικές δικλείδες ασφαλείας για τους πολίτες μας και διευκολύνει τη Διατλαντική Συμφωνία στην καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο Γιούροβα. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ, Χαίρομαι που είμαι και πάλι εδώ για να συζητήσουμε το σημαντικό θέμα της διατλαντικής ροή δεδομένων. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή έχει εργαστεί σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στις διατλαντικές ροές δεδομένων ύστερα από τις αποκαλύψεις Snowden το 2013. Τα κύρια μέτρα λοιπόν αυτά περιλαμβάνουν τον, ε, την υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής ε, μεταρρύθμισης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μια συμφωνία ομπρέλα ε, για τα δεδομένα που ανταλλάσσονται προκειμένου να ε, χρησιμοποιηθούν για την επιβολή του νόμου και την ε, ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Ηνωμένων Πολιτειών για ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων για τις εμπορικές ε, συναλλαγές και τα προσωπικά δεδομένα. Η ασπίδα αυτή έχει ουσιώδη σημασία για τη συνέχιση των διακρατικών ρόλων δεδομένων και εξασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μας και την προσοχή των προσωπικών του δεδομένων. Τη διαπραγματευτήκαμε με τις ΗΠΑ με βάση 13 ε, συστάσεις του Νοεμβρίου του 2013 και δεύτερον οπωσδήποτε των κριτηρίων, βάσει των κριτηρίων που είχε προσδιορίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφαση Σρέμς. Ύστερα από δύο ε, έτη συνομιλιών μπορώ να σας πω ότι έχουμε αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του παλαιού συστήματος του ασφαλούς λιμένα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να συνοψίσω τις κύριες βελτιώσεις. Οι ΗΠΑ καταρχάς οι οποίες λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα από την Ευρώπη θα πρέπει να τηρούν πιο αυστηρούς κανόνες για το πώς θα αξιοποιούν και θα ε, επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες και ε, σχετικά με τη συμμόρφωσή τους η οποία θα παρακολουθείτε από κοντά και προληπτικά από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ. Δεύτερον, ιδιότητα εργοδότες οι οποίοι θα έχουν ε, οι ιδιώτε θα έχουν πρόσβαση σε αριθμό μηχανισμών αποκατάσταση ή ένδικα μέσα για να, για να εξασφαλίσετε ότι κάθε προσπάθεια του για αποκατάσταση των δικαιωμάτων Του θα εξετάζεται και θα αντιμετωπίσετε σωστά. Τρίτον, έχουμε λάβει γραπτέ δεσμεύσει και διαβεβαιώσεις ω προ του περιορισμού και τι ασφαλιστικέ δικλείδε σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα από την, που, χρησιμοποιούν οι αρχέ των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει μόνο δηλαδή την χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων για τον χώρο της ε, εθνικής ασφάλειας. μας έχουν διαβεβαιώσει οι αρχές της ΟΠΑ ότι μια χίδιν συλλογή μπορεί να αξιοποιείται μόνο σε εξαιρετικές ε, περιστάσεις και ότι ακόμη και τότε θα αξιοποιούνται φίλτρα και άλλες τεχνικές οι οποίες θα λεξιτοποιούν το, το συλλεγόμενο όγκο των δεδομένων. Είναι η πρώτη φορά που μας δίδεται μια τέτοια διευκρίνηση και δέσμευση από πλευρά των ΗΠΑ ότι πρόκειται να κάνουν μαζικές ή αδιάκριτες παρακολουθήσεις πολιτών και εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πλαίσιο πολύ πιο ε, στέρεο και στεναρό από ό,τι ήταν το σύστημα του ασφαλούς λιμένα. Τέταρτον, στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας της προσωπικής ζωής και του ιδιωτικού βίου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, η υπηρεσίες των ΗΠΑ θα ε, συστήσουν για πρώτη φορά ένα μηχανισμό ε, διαμεσολαβητή ή ε, εκπροσώπου των πολιτών που θα εξασφαλίζει ότι κάθε είδους προσφυγή ή ένδικο μέσο πολιτών των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα πρόσβασης στα δεδομένα τους αντιμετωπίζεται σε εύθετο χρόνο και πιστεύω ότι αυτό είναι μια άνευ προηγουμένου εξέλιξη και πάλι με πολύ, σε πολύ περιορισμένο βαθμό μπορεί αυτό να συγκριθεί με το, σύστημα του παλαιού, το παλαιό σύστημα του ασφαλούς λιμένα εν τέλει, άπαξ και τεθεί σε εφαρμογή το, το σύστημα αυτό της ασπίδας προσπλασίας του ιδιωτικού βίου, θα παρακολουθείτε διαρκώς, ιδιαίτερα με μια αιτήσια κοινή αναθεώρηση και έκθεση και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα επαληθεύουμε ότι θα υπάρχει σαφής εποπτεία και από κατάσταση και σχετική μηχανισμοί από κατάσταση των δικαιωμάτων και θα, ότι θα λειτουργούν αποτελεσματικά. Έχουμε διατυπώσει σαφείς προϋποθέσεις ε, υπό τις οποίες μπορεί και να άρουμε την απόφαση περί συμμόρφωση, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις από πλευρά των ΗΠΑ. Όπως ξέρετε, η αρχές, οι ανεξάρτητες αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων κατέθεσαν ε, μέσα από το, την ομάδα εργασίας του άρθρου 29, τη γνωμοδότησή τους για την ασπίδα προστασίας του ιδιωτικού βίου, όπου καλωσορίζουν τις θετικές εξελίξεις, αλλά ταυτόχρονα εκφράζουν κάποιες ανησυχίες και συνιστούν περαιτέρω βελτιώσεις αυτές τις πραγματογνωμοσύνες τις λαμβάνουμε υπόψη πολύ σοβαρά. Τώρα δουλεύουμε στα πιο κρίσιμα σημεία και ε, προσαρμόζουμε την απόφαση περί συμμόρφωσης αντίστοιχα. Ε, κάποιες από αυτές τις συστάσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο βέβαια αν συμφωνήσουμε με τις αρχές των ΗΠΑ, πράγμα το οποίο πραγματοποιούμε για διάφορα σημεία και αυτό περιλαμβάνει παραδείγματι τη διευκρίνηση της ανεξαρτησίας και του τρόπου λειτουργίας ε, του διαμεσολαβητή και ε, την πιο σαφή διατύπωση των, του, της αρχής για περιορισμένη διακράτηση προσωπικών δεδομένων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν θέλουμε τα προσωπικά μας δεδομένα και οι αρχές που τα προστατεύουν να ε, κερδίσουν πλήρω πλήρως την εμπιστοσύνη των ιδιωτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Και σε αυτό βέβαια αντιλαμβάνονται και οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι εταίροι μα, ότι είναι πολύ σημαντικέ αυτέ οι διευκρινήσει. Και απαξ και έχουν διευκρινιστεί τα απαραίτητα σημεία και έχουν γίνει βελτιώσει. Θα υποβάλουμε το σχέδιο στα κράτη-μέλη μέσα από την Επιτροπή του άρθρου 31, με στόχο πάντα μέχρι το καλοκαίρι να είναι έτοιμο το πλαίσιο και να λειτουργεί. Και έτσι περνώ στο επόμενο σημαντικό θέμα που σύντομα θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συνένεση τη Συμφωνία ε, ομπρέλας η οποία στοχεύει στην διασφάλιση προστασίας προσωπικών δεδομένων που στο μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την συνεργασία στην ε, τήρηση του νόμου. Η υπογραφή της συμφωνίας αυτής, συμφωνίας ομπρέλας, αναμένεται να λάβει ε, χώρα στην ε, Υπουργική Διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωση Πολιτειών ε, για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών στο Άμστερνταμ στις 2 Ιουνίου. Το Κοινοβούλιο θα κληθεί να δώσει τη συνένεσή του πριν ε, το Συμβούλιο να καταλήξει σε απόφαση για τη συμφωνία αυτή. Ζητώ την υποστήριξη σας για τη συμφωνία Ομπρέλα γιατί θα εξασφαλίσει σαφείς βελτιώσει σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαπιβάζονται στο πλαίσιο της ε, Διατλαντική συνεργασίας για την τήρηση και επιβολή του νόμου σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Όπω γνωρίζετε αυτή η συμφωνία δεν επιτρέπει μεταφορά προσωπικών δεδομένων ούτε αποτελεί απόφαση συμμόρφωση των αντίων ή καλύτερα θα το περιγράψω ε, προσθέτει απαραίτητε διασφαλιστικέ δικλείδε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε υφιστάμενε συμφωνίε για μεταφορά δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση ή κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή όπου αυτέ ε, οι ε, μεταβιβάσει δεδομένων γίνονται με βάση το εθνικό δίκαιο. Πολύ ε, πολλά από αυτά τα μέσα για την τήρηση του νόμου ε, με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε μέχρι τώρα δεν έχουν ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Πρόκειται για ένα status quo το οποίο δυστυχώς υφίσταται και το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει η Συμφωνία Ομπρέλα. Χωρίς τη Συμφωνία Ομπρέλα αυτή η μη ικανοποιητική κατάσταση θα μπορούσε να συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα και όποτε διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα ε, Αμερικανών υπηκόων στην Ευρώπη, θα μπορούν και αυτοί να έχουν ένα υψηλό επίπεδο προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπω ορίζουν οι δικοί μα κανόνε, είτε πρόκειται για το ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε πρόκειται για το εθνικό δίκαιο. Και ω εκ τούτου η συμφωνία Ομπρέλα έχει σαν στόχο και να, να αποκαταστήσει τι ανισορροπίε, αλλά και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στι διατλαντικέ μεταφορέ δεδομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Ε, για δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριο Φως. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Υπουργέ, κυρία Πίτροπε. Χρειάζεται επιγόντως μία διάδοχη κατάσταση του Safe ε, Harbor. Το θέμα αυτό σας ε, προστασίας ιδιωτικής ζωής είναι βελτίωση. Η πολιτική διαμάχη εδώ έχει να κάνει με τη ρήτρα εκπνοής. Sunset Close και συμφωνήσαμε κατά πλειοψηφία να μην υιοθετηθεί τέτοια, άρα περιμένω και από τους συναδέλφους ε, των φιλελευθέρων και των σοσιαλιστών και δημοκρατών ε, να μην υποστηρίξουν τις τροπολογίες των πρασίνων και ε, της ενωτικής αριστεράς. Αλλά μια τέτοια ρήτρα δεν χρειάζεται καθόλου κατά την άποψή μου, διότι έχουμε έναν ισχυρό ετήσιο μηχανισμό εποπτείας που μπορεί σε μόνη βάση να κάνει στην άκρη κάποια υπόλοιπα. Είναι ένα στιβαρό πλαίσιο διαρκές και μια τέτοια ρήτρα θα ήταν άχρηστη και περίτη εάν ε, υπάρχει πραγματικά ένας τέτοιος μηχανισμός που να λειτουργεί. Για να δούμε λοιπόν, να περιμένουμε ε, αν θα λειτουργήσει πριν το σταματήσουμε και πάλι. Αυτό που είναι το θέμα εδώ είναι η καχυποψία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δυσπιστεί ότι μπορεί να παρακολουθήσει και να πλαισιώσει αυτή τη διαδικασία, αλλά νομίζω ότι έμαθε το μάθημά τη πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ε, απαιτήσει για μια σπίδα προστασία ιδιωτική ζωή είναι και πολιτικά γελία κατά την άποψή μου. Από εκεί και πέρα πώ θα κρίνει και ποιο θα κρίνει αν αρκεί αυτή η ασπίδα ή όχι. Είμαστε λίγο ανερμάτιστοι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μεγαλύτερες και οι νεοφυείς θα πρέπει να έχουν μια ασφάλεια δικαίου, να ξέρουν σε ποιο πλαίσιο κινούνται ε, για την ε, διατλαντική ε, διαβίβαση δεδομένων. Εμείς θα υποστηρίζαμε αυτή την ασπίδα. Αν όμως περάσουν οι συγκεκριμένες τροπολογίες, το ΕΛΚΑ την καταψηφίσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριος Βάιντεν Χέλτσαρ για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε. Το θέμα αυτό τώρα μας απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επί της ουσίας διαφωνούμε. Ε, συζητούσαμε πάντα και συγκρουόμαστε για το safe harbor με διάφορους τρόπους και υπήρξε και ανασφάλεια που ε, ανασφάλεια δικαίου που ήρθε να λυθεί από την προσφυγή ενός πολίτη. Και αυτή η απόφαση ΣΡΕΜΣ έχει ε, μπει πλέον στην ιστορία, ανήκει στα χρονικά. Ε, το Privacy Shield, η ασπίδα ε, προστασίας, είναι μια πρώτη απόπειρα να λυθεί το πρόβλημα. Το Φεβρουάριο μας παρουσιάσατε τις γενικές αδρές γραμμές. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος και με την ομολογία μπορέσαμε να λύσουμε κάποια πράγματα με τους Αμερικανούς εταίρους. Παραμένει όμως η κατάσταση ε, επισφαλής, ανασφάλεια επικρατεί. Δεν έχουμε πια και την σοπερσαφήνεια, δεν είναι κρυστάλλινα τα πράγματα, άρα υπάρχει κινδυνός να καταλήξει και άλλη υπόθεση στο δικαστήριο ε, και αυτό για το δικό μας κύρος ως νομοθετών και εκτελεστικής εξουσίας δεν θα ήταν ε, απαραίτητα θετικό. Ούτε για την οικονομία είναι αυτό θετικό. Την περασμένη εβδομάδα η Επιτροπή Ελευθεριών ε, μετέβημε στι ΗΠΑ και εκεί είδαμε ότι υπήρξε μεγάλη κατανόηση για την ευρωπαϊκή ε, πλευρά και θέση και έχουν και προθυμία να ανταποκριθούν στη δικαστική απόφαση. Αυτό ισχύει και για τις κρατικές δομές αλλά και για την ε, η οικονομία των δεδομένων, τις εταιρείε που χειρίζονται τα δεδομένα, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μεγαλύτερη πρόοδο. Καλό είναι να ορίζουμε κάποια κριτήρια. Λοιπόν, χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, σαφήνεια. Τι θα πει γραπτή ε, διαβεβαίωση. Αυτό έχει κάποιο νομικό χαρακτήρα και ισχύει. Και το judicial redress που είναι τόσο σημαντικό δικαστική ε, αποκατάσταση θα πρέπει να ξέρουμε τι είναι και να μην ισχύει μόνο για πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μας ικανοποιεί αυτή η διατύπωση γιατί έχουμε και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ευρώπη και προστατεύονται από το χάρτη των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτές οι βεβαιότητες θα πρέπει να ε, απομακρυθούν Καλό είναι που κάναμε αυτή την προσπάθεια από κοινού. Μόνοι μα δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Παρακαλώ όμω λύστε τα αυτά τα θέματα που εκκρεμούν ακόμα και τα σαφή. Αλλιώ θα ξανανοίξει η συζήτηση κτλ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο. Η κυρία Στέβεν για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι η διατλαντική μεταφορά δεδομένων είναι πάρα πολύ απαραίτητη για την οικονομία, για το εμπόριο και την ασφάλεια. Ε, με τη νέα σπίδα τώρα έχουμε μια νέα μορφή προστασίας. Είναι ένα μεγάλο βήμα πραγματικά προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα δικαιώματα και η προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών κατά τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ κάνει άλμα υπάρχουν κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεωρούν ότι απλώς ε, θα αρκούσε να ε, μεταφέρουμε το Ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασία. Μα οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι και ανεξάρτητο κράτο και σημαντικό εταίρο. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι δεν είναι μέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Ηνωμένε Πολιτείε και έχουν δική του αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Οι νέοι κανόνε θα πρέπει ε, να μπορούν να αντέχουν στη δοκιμή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών ε, Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον για να ε, μπορούν οι εταιρείε να δουλεύουν σε ένα πλαίσιο ασφαλές. Η ευρωπαϊκή οικονομία θα πρέπει να ε, προστατεύεται αλλά και η ιδιωτική ζωή των πολιτών, οπότε θα πρέπει το συντομότερο το Privacy Shield να γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέλτ για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να ξεκινήσω απειχώντα τα τελευταία λόγια τη κυρία Στίβεν, ότι επιθυμούμε να έχουμε ε, μια ε, επιχειρησιακή ασπίδα ε, προστασία όσο γίνεται πιο σύντομα. Το πρόβλημα είναι όμω ότι δεν θα είναι επιχειρησιακή. και βρισκόμαστε εδώ χάρη στον στον Σρέμσε που είχε το θάρρος να αγωνιστεί στο δικαστήριο εδώ και χρόνια και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Ευρωπαίου πολίτη. Γιατί εδώ επανειλημμένα ζητήσαμε την απόρριψη του, του, του ασφαλούς λιμένα. Ένας αυστριακός φοιτητής εξασφάλισε ε, την ε, απόφαση αυτή. Και δεν είμαι καθόλου πεπισμένη ότι οι γραπτές αυτές διαβεβαιώσεις ή, ή ο διαμεσολαβητής ή με αναθεώρηση κτλ. θα τα καταφέρουν. Η ομάδα εργασίας το EDPS και διάφοροι νομικοί εμπειρογνώμονε λένε ότι δεν θα λειτουργήσει. Γιατί πρέπει να λέμε τα ίδια και να κάνουμε τα ίδια λάθη ξανα και ξαναμανά. Έχουμε ευθύνη και καθήκον να κάνουμε νομοθεσία ποιότητα Και έχω την εντύπωση ότι εδώ η Επιτροπή είναι έτοιμη να λάβει μια απόφαση που δεν πρόκειται να σταθεί σε καμία περίπτωση στο δικαστήριο. Εδώ εγώ δεν θέλω να κάνω πολιτικέ συμβιβασμό. σω θα μπορούσα να συμφωνήσω με τον κύριο Βόλσο, ίσως όχι. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση. Ε, μόνο ένας γνώμονας πρέπει να υπάρχει. Είναι ναι ή όχι ε, αδιάβλητο στην απόφαση ΣΡΕΜ. Δεν είμαι βέβαιη ότι είναι. Πρόκειται για βελτίωση, ναι. Είναι ένα βήμα μπροστά. Είμαι ευτυχή που η Κομισιόν θέλει να συζητήσει περαιτέρω προσαρμογέ, αλλά τελικά Πρόκειται για την πρόσβαση των ΗΠΑ σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων ε, καταναλωτών και εκείνοι έχουν λοιπόν συμφέρον να κινηθούν. Τέλο, δεν είπαμε τίποτα για τη συμφωνία ομπρέλα στο ψήφισμα, θα επανέλθουμε, αλλά πραγματικά θα ήθελα τα εξή δύο πράγματα. Καταρχά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν να μιλήσουμε για συγκατάθεση οτιδήποτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποχαρακτηρίσει την απάντηση που έδωσε στην ΛΥΜΠΕ για το νομικό καθεστώς και το, πεδίο, ε, το εύρος εφαρμογή της ε, Συμφωνίας Ομπρέλα. Δώστε μας αυτή την πληροφορία. Αυτό είναι απλά μια νομική αξιολόγηση, εκτίμηση. Πόσο απόρριτη μπορεί να είναι. Και δεύτερον, η Κομισιόν ίδια έχει δηλώσει ότι η αφαίρεση των ε, ε, εξαιρέσεων για την ιδιωτική ζωή στη ΣΥΠΑ ε, είναι προϋπόθεση. Δεν πρόκειται να αφαιρεθούν αυτές οι εξαιρέσεις. Μπορεί λοιπόν κάποιος να με εξηγήσει πώς γίνεται ε, ρεαλιστικά να αναμένουμε ότι αυτή η συμφωνία ομπρέλα θα εφαρμοστεί. Για πείτε μου, για εξηγήστε μου παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Εάνστα έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι. Μπορούμε να το ονομάσουμε και privacy shield, άμα θέλετε. Αλλά το θέμα είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα των 500 εκατομμυρίων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά πρέπει να τα προστατέψουμε και σε σχέση με τα, προσω... με τα ιδιωτικά συμφέροντα. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε μόνο ένα... Ε, μία κατά τα φαινόμενα προστασία. Χρειάζεται μια ουσιαστική προστασία. Και Βεβαίω μπορεί μεγάλη εδώ ε, συνεργασία και συμμαχία να υποστηρίζει αυτή την ε, λύση, αλλά ούτε καν ένα sunset clause δεν μπόρεσε να δεχθεί να εισαχθεί στη συμφωνία αυτή η ομπρέλα. Και αυτή η νέα συμφωνία δεν έχει καν χαρακτήρα συνθήκης. Δεν έχει νομοθετικό υπόβαθρο. Ο Τζον Κέρι μάλιστα λέει ότι δεν θα μπορεί ο Ombudsman, τον οποίο υποτίθεται ότι προσφέρουμε στους Ευρωπαίους πολίτες, να επικυρώνει ή να ακυρώνει αποφάσεις. Τι είδους Ombudsman θα είναι αυτός λοιπόν. Και εδώ, όπως είπα, κυρίες και κύριοι, διακυβεύονται τα δικαιώματα 500 εκατομμυρίων πολιτών. Δεν μπορούμε να τα θεσιάσουμε στο βωμό ενός πραγματικού μεγάλου αδελφού. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Ευχαριστώ πολύ. Άλμπρεχτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. κύριε Επίτροπε, δουλέψατε μας με την ομάδα σας σκληρά για να καταλήξετε στο αποτέλεσμα αυτό για την ασπίδα προστασίας του ιδιωτικού βίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτειών και για τη Συμφωνία Ομπρέλα. Και όντως σημειώθηκε πρόοδος. Αλλά είμαστε και ειλικρινείς. Στα θέματα προστασίας του ιδιωτικού βίου στη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένων Πολιτειών πραγματική βελτίωση σε σχέση με το σύστημα του ασφαλού λιμένα δεν υπάρχει γιατί δεν άλλαξε το νομικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό ακριβώ ήταν που έχει επισημάνει ε, και στη λιτεύση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου ότι δεν προσφέρει το νομικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών ε, ε, ασφαλή προστασία. Πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό και εφόσον και από τη στιγμή που καταγράφουμε όλες τις επικρίσεις και όλα τα ελλείμματα του συστήματος αυτού, πώς είναι δυνατόν να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται πάνω από τη διαπραγμάτευση στο μέλλον, χρειάζεται να ξανανοίξουμε τα θέματα αυτά στη διαπραγμάτευση γιατί δεν έχουμε φτάσει στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Δεν, λέμε αυτό, αλλά λέμε όχι, τα έχουμε καταφέρει όλα, βάλαμε μερικές δυσφαλιστικές δικλείδες, ψηφίζουμε και βλέπουμε στο μέλλον τι θα γίνει και μπορεί και το δικαστήριο κάποια στιγμή να ε, καταρρύψει το σύστημα αυτό. Ας είμαστε ειλικρινείς λοιπόν. Η μόνη ειλικρινή στιγμή στη συζήτηση αυτή θα ήταν να οριστεί μια ρήτρα εκπνοής, μια sunset clause και να ανατραπεί η κατάσταση, η συμφωνία αυτή. με που δεν μπορούν να δεχθούν τη λύση αυτή οι λοιπές ομάδες. Και για να είμαστε και ακόμη πιο ρεαλιστικοί εμείς, ε, ζητήσαμε με μια νέα τροπολογία τέσσερα χρόνια διάρκειας, που έτσι θα, θα επέτρεπε σε μια νέα κυβέρνηση ΗΠΑ να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό σας παρακαλώ όλοι να δεχτείτε την τροπολογία μας. Ευχαριστώ πολύ. Μπέγκιν ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, εδώ σε ποιον ανήκουν ε, τα προσωπικά δεδομένα που οι Ευρωπαίοι διαβιβάζουν ε, στη ΣΥΠΑ με το στο Google, Instagram και ούτω καθεξής. Τι εγγύηση έχουν ότι η περιοδική του ζωή δεν θα παραβιάζεται διαρκώ καμία. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι ελεύθερη να ε, διαχειρίζεται τα στοιχεία των ξένων όπως θέλει και επίση οι μυστικές υπηρεσίες μπορούν να τα χρησιμοποιούν. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι ένα ε, αγαθό ανταλλάξιμο είναι η ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και το δικαστήριο το είπε αυτό ρητά. Εγώ θυμάμαι ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό τα τηλέφωνα αυτού του κοινοβουλίου τα mail μας, ακόμα και τα κινητά των βουλευτών κατασκοπεύονταν στους Αμερικανούς. Αυτό έχω να πω για την ιδιωτική ζωή και η συμφωνία που, θέλουμε να υπογρα... που θέλει η Κομισιόν να υπογράψει δεν προβλέπει καμία δεσμευτική πρόταση. Είναι προσβολή στην απόφαση του δικαστηρίου και στις χιλιάδες πολιτών που εμποστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατέψει την ιδιωτικότητά τους. Αλλά η Κομισιόν δεν θέλει προβλήματα για το TTIP που θα αυξήσει την ε, διατλαντική ροή δεδομένων. Ρωτώ, συνάδελφοι, αυτή είναι η όρη που του οποίου θα υπογράψετε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ κύριο Επιτίδιος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα από του μεγαλύτερου κινδύνου που έχει δημιουργήσει στον σύγχρονο άνθρωπο η ραγδαία εξέλιξη τη τεχνολογία είναι η υποκλοπή των προσωπικών δεδομένων από τι ιστοσελίδε κοινωνική δικτυώσεω και η επεξεργασία του από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ιδιαίτερα στι ηνωμένε πολιτείε ο κίνδυνο αυτό έχει λάβει τεράστιε διαστάσει διότι η ίδια η νομοθεσία επιτρέπει στι υπηρεσίε πληροφοριών τη γνωστή μα cia και την υπηρεσία ε, εθνική ασφαλεία την nsa να συλλέγουν να επεξεργάζονται και να διατηρούν τέτοιου είδου πληροφορίε πολλέ φορέ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο τη πενταετία μάλιστα στο όνομα ε, του εθνικού συμφέροντος των ηπα οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να συλλέγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες όχι μόνο αμερικανών αλλά και υπηκόων άλλων κρατών στα ίδια τους τα κράτη μάλιστα. με αυτόν τον τρόπο όμως παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα καταστρατηγείται το δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων δυσχεραίνεται η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού εμπορίου ε, και επιπλέον δημιουργείται μια νομική αβεβαιότητα σε επιχειρήσει και φυσικά πρόσωπα. γι' αυτό το λόγο η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα ούτω ώστε στο διάλογο με τι ΗΠΑ για τη ρύθμιση των όρων τη ασπίδα προστασία τη ιδιωτικής ζωής να επέρθουν οι βελτιώσει εκείνες που θα εξασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων των ευρωπαίων πολιτών που έχουν εμπορικέ δραστηριότητε με τις ΗΠΑ. Πολιτείε. Δέχεστε μπλε κάρτα. Από τον κύριο Σάνι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη συζήτηση αυτή πολύ συχνά ακούσαμε ότι η μεταφορά δεδομένων και ανταλλαγή δεδομένων δεν έχει να κάνει μόνο με το εμπόριο. Μπορείτε να επαναλάβετε παρακαλώ. Ευχαριστώ ε, Πρόεδρε. Έλεγα λοιπόν, αρχίζω ξανά, ότι ε, στη σημερινή συζήτηση επανειλημμένα ακούσαμε ότι η προστασία δεδομένων δεν έχει να κάνει μόνο με το εμπόριο, αλλά ε, το θέμα που μας απασχολεί δεν είναι εμπορικό ζήτημα, δεν είναι κανονικό εμπόριο και ξέρουμε που μπορούμε να οδηγηθούμε όταν χρησιμοποιούν τα δεδομένα μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις σε περίπτωση καταχρήσεων. Ε, Βεβαίω, πρέπει να επιβληθούν κυρώσει, όμω προηγουμένω θα πρέπει να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θα αποτρέψουν να εκτραπούμε προ αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν ε, απαιτούνται και τα δύο και προσπάθεια να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο αλλά όταν όμως γίνει παραβίαση προσωπικών δεδομένων ναι πρέπει να έχουμε κυρώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λέναρτς για μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε διατλαντική ροή δεδομένων είναι τεράστια στον κόσμο. 15 τεραμπάιτ το δευτερόλεπτο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία μας, για την κοινωνία μας που ψηφιοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς και εκεί βρίσκεται και μια ελπίδα για το μέλλον. Ε, υπάρχει όμως ένα νομικό κενό και μια ανασφάλεια που υπήρχε στο παρελθόν. Ε, είναι 5.000 εταιρείε που χρησιμοποιούν ε, τους πρώοι του Safe Harbor και κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε τέτοιες καταστάσεις. Ε, τώρα καλούμαστε με ένα σπάρο να σκοτώσουμε δύο τριγώνια. Προστασία των δεδομένων, βέβαια των πολιτών από τη μια και από την άλλη που είναι επίσης σημαντικό, ασφάλεια δικαίου για τις εταιρείες που κάνουν χρήση αυτής της ε, ρύθμισης. Χαίρομαι με τη δουλειά που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόοδος προέρχεται και από ε, πολλές κατευθύνσεις και την έχουν ε, σήμερα εκθιάσει πολλοί συνάδελφοι. Υπάρχει ομάδα εργασία ε, του άρθρου 29 που θα πρέπει να ε, το δει τι επόμενες εβδομάδες. Εμείς τη ζητάμε. Φροντίστε φέτος το καλοκαίρι να λήξει αυτή η υπόθεση, να υπάρχει μια ασπίδα προστασίας ε, της ιδιωτικής ζωής, να αισθάνονται οι πολίτες άνετα, αλλά να προχωρήσουν και επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε η κυρία Γκόμε για δυόμιση λεπτά. Πήγα στην αντιπροσωπεία με τη Λίμπε στη ΣΥΠΑ. Είχαμε, ήρθαμε σε επαφή με διάφορους συνομιλητές και εκπροσώπους των μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις ροές δεδομένων ε, και μάθαμε ότι πρόκειται για ένα πλαίσιο σφαιρικό ε, για συμφωνία χωρίς ε, προηγούμενο, μέσω του οποίου θα μπορούσαμε να προσφέρουμε υπηρεσίες σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και περισσότερη δικαστική ασφάλεια. Αυτές οι παράμετροι διέπουν αυτή τη συμφωνία που προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό σε αυτή την ε, ψηφιακή εποχή που δεν είναι μόνο ψηφιακή οικονομία να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στις διατλαντικές ανταλλαγές στοιχείων και να εγγυηθούμε στις επιχειρήσεις και στους πολίτες ε, νομική ασφάλεια με ένα ε, στεναρό σύστημα για να να μην, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μπορούν μάλλον να χρησιμοποιηθούν για τις ε, ποινικές ε, έρευνες. Ε, Θα πρέπει να γίνει αυτή η διαπραγμάτευση και η συνομιλία, η, η, γιατί υπάρχουν ακόμα επιφυλάξεις όσον αφορά την συμβατότητα με το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο και με βασικά θεμελιώδη, θεμελιώδη νομολογία του ΔΕΚ. Ε, υπάρχουν ε, οδοί προσφυγής, αλλά είναι πολύ περίπλοκες για τον κοινό πολίτη. Θα πρέπει επίσης να μπορούν... Ε, να καλύπτονται δε και οι μη Ευρωπαίοι πολίτε που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τελείω υπάρχει διάκριση σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή ε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όπως και οι Αμερικανοί συνομιλητές μας έχουμε επιφυλάξει όσον αφορά το γεγονός ότι ο πάροχος δεν έχει ένα συγκεκριμένο καθεστώς σε σχέση με τους διοικητικούς μηχανισμούς. Επιτρέπεται δε η συλλογή δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα ε, αντίθετα με τις αρχές της επικουρικότητα και της αναλογικότητας που εντάσσονται στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να προστατευτούν ε, τα δικαιώματα των Αμερικανών και Ευρωπαϊκών Ευρωπαίων πολιτών μέσω ε, σωστής νομοθεσίας. Θα πρέπει λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο να εκφράσει τις επιφυλάξεις του και να ζητήσει από την Κομισιόν και από τη ΣΥΠΑ να επιβάλλει αυτές τις ε, ε, συνομιλίες στην ομάδα εργασίας 29 να τηρηθούν οι κανονισμοί σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να γίνει σεβαστή απόφαση ΣΡΕΜΣΕ και επίσης να προστατευτούν τα βασικά δικαιώματα των ε, πολιτών. Ευχαριστώ. Κυρία, Κυρία ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη υιοθετήσει μια σειρά συμφωνιών για την προστασία προσωπικών δεδομένων, για την, για την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μάλλον και για την ε, δίωξη των ε, τρομοκρατών που απειλούν ε, την ασφαλειά μας. Θα διευκολυνθεί ασφαλώς το οικονομικό περιβάλλον με την ανταλλαγή των δεδομένων οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με τις Ηνωμένε Πολιτείες μπορεί όμως να επιβαρυνθούν με σαφή γραφειοκρατικό φόρτο ο ιδιωτικός βίος, ε, οι ελευθερίες των πολιτών και έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να γίνουν σεβαστά και πρέπει να αποτραπούν επιθέσεις εις βάρος των δικαιωμάτων και παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών. Πρέπει λοιπόν το χειρότερο δυνατό να υψωθεί αυτή η ασπίδα προστασίας για τον ιδιωτικό βίο των πολιτών, να παρακολουθηθεί και να αξιολογηθεί ο τρόπος εφαρμογής της, που πιστεύω ότι είναι απαραίτητη. Α ξεκινήσει όμω η εφαρμογή και μετά θα γίνει η αξιολόγηση. Τι άλλο δεν πρόκειται να έχουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Μπάτν ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ψηφίσουμε το... Έχουμε το ψήφισμα αυτό να ψηφίσουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση την διαβίβαση προσωπικών δεδομένων των πολιτών και έχει σαν στόχο, λέει, το είναι ισχυρότερη προστασία των δεδομένων και των προσωπικού βίου. Οι ιδιωτικέ επιχειρήσεις βέβαια έχουν και έναν τρόπο με τον οποίο προσδιορίζουν στις συμφωνίες τους το, τη χρήση των δεδομένων των πολιτών ωστόσο κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει στη σχέση ενός πολίτη με ένα κράτος. Δεν υπάρχει ζήτημα συνένεσης. Ε, ένα κράτος, μια κυβέρνηση πρέπει να χρησιμοποιεί τα δεδομένα με κάθε σεβασμό και προσοχή. Υπάρχουν ανησυχίες βεβαίως προς την αξιοποίηση προσωπικών δεδομένων από τις ΗΠΑ που έχουν μειώσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δικών του ήδη πολιτών με νομοθετήματα όπως το Patriot Act που ποτέ δεν, οδηγεί, δεν μπορούσαν να αποκαταστήσουν τα δικαιώματα και γι' αυτό εμείς θα καταψηφίσουμε το ψήφισμα. Γιατί η αδίποτε νομοθεσία πρέπει να παραμένει αρμοδιότητα και στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους εθνικού και κυρίαρχου. Ευχαριστώ πολύ. Νίμπλερ, 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, κύριε Προεδρεύον του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι θέλουμε τη διαβίβαση των διατλαντικά των δεδομένων ή όχι. Εγώ νομίζω ότι τα χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε να, υπάρχουν αυτέ οι ροέ διατλαντικών προσωπικών δεδομένων, αλλά ταυτόχρονα και την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίε δεν είναι σε θέση να ε, διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους ε, μέσα από συμβάσεις προσχωρήσεως ή άλλες μαζικές συμβάσεις και άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία. Είναι πολύ σκληρή η δουλειά που έκανε η Επιτροπή με τις διαπραγματεύσεις της επί πολλούς μήνες και νομίζω ότι συνιστά σημαντικό, ε, σημαντική βαλτίωση η τωρινή συμφωνία σε σχέση με την προηγούμενη του ασφαλούς λιμένα. Η ασπίδα προστασίας εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων, έχει διατάξεις και διατυπώσεις για πιο προσεκτική χρήση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και στις ΗΠΑ. Βέβαια, εν τέλει, από την πρακτική υλοποίηση της συμφωνίας θα κριθεί η επιτυχία της. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να γίνονται και οι αιτήσει αξιολογήσεις της εφαρμογής της και όχι μόνο οι αξιολογήσεις, αλλά αν τυχόν και προκύψει ακόμη και η εντύπωση πως δεν είναι αρκετά προσεκτική η διαχείριση των δεδομένων από τις ΗΠΑ, θα πρέπει να αρθεί το αξιόπιστο της συμφωνίας. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια καλή λύση. Υπάρχει δυνατότητα της βελτίωσης χάρη στην ομάδα του άρθρου 29, είτε τώρα είτε σε μια μεταγενέστερη φάση αξιολόγησης και νομίζω ότι είναι μια καλή συμφωνία για μας και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Μακλάρκιν, ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να αναγνωρίσουμε τα βήματα προόδου που σημείωσαν οι Αμερικανοί εταίροι μας τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση της προστασίας ροών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ, ανταποκρινόμενοι απευθείας στις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί ιδιαίτερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Κογκρέσο και η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχουν προχωρήσει 24 τουλάχιστον νομοθετήματα καινούρια, μεταρρυθμίσεις όπως το Privacy Shield και άλλα αντίστοιχα και όπως και άλλοι συναδελφοί θεωρώ ότι πρόκειται και μια ευκαιρία ε, η συμφωνία που έχουμε με την ασπίδα προστασίας, εκτός για, για την προστασία των δεδομένων των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων και πρέπει αντίστοιχα να ε, προχωρήσουμε και σε συμφωνίες όπως η ΤΕΖΑ, όπως η TTIP. Δηλαδή να έχουμε συμφωνίες οι οποίες θα είναι αμοιβαία επωφελής και για τις δύο πλευρές. Έχουμε να κάνουμε 3 δισεκατομμύρια ε, αμερικανικά δολάρια σε συναλλαγές και χρειάζεται και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και οι δυνατότητες για άσκηση ενδικών μέσων από τους πολίτες για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φωνστόρχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Συζητούμε εδώ τώρα για τη ροή δεδομένων, ανταλλαγή δεδομένων με τη ΣΥΠΑ και για την προστασία των δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται αυτό τον καιρό μια νέα συμφωνία προς την κατεύθυνση αυτή ακριβώς διότι μεσολάβησε δικαστική απόφαση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάστηκε να προσφύγει ένα πολίτης γιατί διαπίστωσε ότι η προστασία των δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δεδομένη. Εξού και η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανησυχούμε βαθύτατα, έχουμε θορυβηθεί. Ε, σημείωσα όλα αυτά που είπατε, αλλά δεν με κάνουν αισιόδοξη μας λέτε ότι δεσμεύονται οι Ηνωμένε Πολιτείε, μας διαβεβαιώνουν, μας τάζουν, ε, λαγούς με πετραχίλια. Ωραία. Ε, αν δεν έχουμε συμφωνία τελικά που να ε, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να προσφεύγουν στα δικαστήρια και να επιβάλλεται η απόφαση, δεν θα έχει περισσότερη αξία συμφωνία αυτή από αυτό το στυλό που κρατάω στα χέρια μου. Ευχαριστώ. Μπόνι, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ και σας και το επιτελείο σας ε, για την εξαιρετική δουλειά. Και τώρα νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος ε, της ιστορίας αυτής που σημαίνει ότι θα έρθει αυτή η ασπίδα προστασίας στην ζωής. Όλοι ξέρουμε τι σημασία έχει ε, αυτός ο κλάδος τη ροής δεδομένων στη σύγχρονη οικονομία. Χρειάζεται σωστή λύση για όλους και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν λιγότερες δυνατότητες και νομικές και επενδυτικές ε, και ε, που θα επωφεληθούν από μια τέτοια συμφωνία. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε την ασπίδα προστασίας για να ε, αυξηθεί η σημερινή ψηφιακή οικονομία. Είναι καλή προσέγγιση αυτή θα πρέπει με τη συμφωνία να επανέλθει η εμπιστοσύνη κατέρθεν του Ατλαντικού. Η πρόταση εισάγει πολλές βελτιώσεις στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων μεταξύ άλλων, ενισχύει ε, την προστασία ε, των δεδομένων με τις αντίστοιχες αρχές στα κράτη-μέλη, Υπάρχουν ένδεικα μέσα που ενισχύονται για τους πολίτες και εκείνους που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργείται και μια ειδική αρχή διαμεσολάβηση Ombudsman. Αυτά, επαναλαμβάνω, έχει σημασία να εφαρμόζονται κατέρωθεν του Ατλαντικού και να αλλάξει και η νομοθεσία αλλά και η νοοτροπία. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα μέσα είναι στη διάθεση των πολιτών της Ένωσης και το κατοίκων της Ένωσης και ότι θα υπάρχει και μια τακτική αναθεώρηση και ο επόπτης προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει το ρόλο του να παίξει και διάφορες εθνικές αρχές. Ο κύριος Γιούζ Αντζουτόφσκι για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ε, για τη συμφωνία αυτή σχετικά με τη ροή δεδομένων από την Ευρώπη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το αντίστοιχο. Είναι ένας παραδοσιακός εταίρος μας, είπα και καλό είναι να κάνουμε αυτή τη συζήτηση στα πλαίσια της αμοιβαία εμπιστοσύνης και όχι αμοιβαία καχυποψίας. Χαίρομαι που βλέπω τις ε, σημερινές προτάσεις για την προσφυγή στη δικαιοσύνη και τη δικαστική αποκατάσταση Θέλω πραγματικά να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων και να εξασφαλίζεται από τη συμφωνία. Θα πρέπει να είμαστε και λογικοί όμως. Καμιά φορά έχω την αίσθηση αυτό το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ερμηνεύεται με τρόπο καταχρηστικό που αντιτίθεται ε, στη συμπεριφορά που έχουμε για άλλα αγαθά. Στα θέματα της ασφάλειας δεν πρέπει να είμαστε τόσο περιοριστικοί γιατί πρέπει να προστατεύσουμε και τους πολίτες μας, όχι μόνο τα δεδομένα τους. Ωραία, πάμε στη διαδικασία Catch the Eye τώρα. Ο κύριος Καπούτο. Σε προηγούμενες ε, παρεμβάσει ακούσαμε πόσο σημαντική είναι η απόφαση του ΔΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 2015. Οι νέε συνομιλίες φαίνεται ε, και η νέα πρόταση συμφωνίας φαίνεται να ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόκληση ε, ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν οι ροές δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς αλλά το εμπόριο ή ε, ε, μάλλον ε, στην συλλογή χίδιν ιδιωτικών στοιχείων έχουν ήδη υπάρξει προβλήματα παλιότερα όμως με τη ΣΥΠΑ και θα είναι δύσκολο να τηρηθούν οι διάφορες υποχρεώσεις όσον αφορά την ιδιωτική ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και τη τήρηση αυτών των υποχρεώσεων. Όμως θα πρέπει να δούμε ποιες διαδικασίες προσφυγής θα περιλαμβάνονται σε αυτή τη συμφωνία που είναι πραγματικά αποτελεσματικές. Σε αυτές τις τεράστιες όγκους στοιχείων είναι αδύνατο να γίνει χώρο όριος έλεγχος και σε περίπτωση παραβίασης θα πρέπει να τονίζεται ο ρόλος της Κομισιόν που εύχομαι δεν θα φτάνει μόνο μέχρι το ΔΕΚ. Ευχαριστώ κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδης δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κάθε μέτρο προκειμένου να μην παραβιάζονται όσον αφορά τι διατλαντικέ ροέ δεδομένων η ευρωπαϊκή ένωση και οι ηνωμένε πολιτείε έχουν υπογράψει συμφωνία για την προστασία τη ιδιωτικότητα και την ασφάλεια του δικαίου για τι επιχειρήσει σε περίπτωση που υπάρχει μεταβίβαση δεδομένων από την ένωση στι ηπα. βέβαια όπω ορίζεται στο πλαίσιο τη νέα ρύθμιση οι δημόσιε αρχέ των ηπα υποτίθεται ότι θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και θα το πράττουν αυτό υποτίθεται υπό περιορισμού και με την επίβλεψη ούτω ώστε να μην υπάρχει γενικευμένη πρόσβαση παράλληλα οι ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν διεξαγωγή έρευνας ή να υποβάλουν καταγγελία σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών τους δεδομένων. ωστόσο είναι αναγκαίο να συγκεκριμενοποιηθούν οι περιπτώσεις πρόσβασης των δημόσιων αρχών των ηπα σε προσωπικά δεδομένα και να επιτευχθεί ισορροπία ασφάλειας και ελευθερίας. η προστασία των δεδομένων σε κάθε διατλαντική ροή θα πρέπει να προστατεύεται και να μην υποτάσσεται στις επιδιώξεις των υπηρεσιών ασφαλείας των ηνωμένων ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λόπε Αγγιλάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλό θα ήτανε να μην έχουμε ροές δεδομένων διατλαντικές. Όχι το κοινοβούλιο οφείλει να αντισταθεί, πρέπει και, μπορεί, όχι βέβαια και είναι και μαζική η μεταφορά, αλλά θα πρέπει να απαιτήσουμε αυτή η ροή δεδομένων να ρυθμίζεται από το δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δουλειά τη την έκανε. Προσπάθησε να συμφωνήσει να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ μία σπίδα προστασίας, που δεν είναι ουρανοκατέβατη γιατί έπεσε ράβδο από το δικαστήριο ε, με την κατάργηση του Safe Haven, του ασφαλούς λιμένα, στην περίφημη υπόθεση ΣΡΕΜΣ και το προδικαστικό ερώτημα. Ωστόσο παραμένουν οι αφιβολίες και θα πρέπει ε, να επαγρυπνούμε για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η νέα συμφωνία και πώς συνάδει με το χάρτη θεμελιτών δικαιωμάτων. Και εδώ αποκτά τεράστια σημασία η ρήτρα της αιτήσιας αναθεώρησης, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβλέπει ε, την τήρηση ε, της συμφωνίας και υπάρχει μια εποπτεία που έχει προσφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα πρέπει να έρθει άλλη μια τέτοια απόφαση κατηγορηματική και ακυρωτική της συμφωνίας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ. Οποιαδήποτε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θεωρούνται ως βάση ε, για να κάθε φορά να πάρει ένωση αρμοδιότητες των κρατών. Ε, σκεπτόμενοι αυτό το γεγονός, ε, είχα αμφιβολίες. Όμως εδώ πρόκειται για μια, ένα πεπαλαιωμένο κανονισμό που δεν παρέχει το ψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Η ασπίδα προστασίας των δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων, δεδομένων δίνει κάποιες εγγύησεις για το σεβασμό των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών ε, πέρα από τον Ατλαντικό και ο Μεσολαβητής. Ε, επίσης είναι πολύ σημαντικός καθώς και η εισαγωγή μιας υποχρεωτικής ε, ε, προθεσμία 45 ημερών για την εξέταση των ε, καταγγελιών των πολιτών. Οι πολίτες θα καλωσορίσουν, ελπίζω, το γεγονός ότι για πρώτη φορά θα εισαχθούν ε, σαφείς περιορισμοί προς τις, ευρωπα... στις αμερικανικές εταιρείες για την πρόσβαση τους στα δεδομένα και έχει, σημαντική, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και την καλωσορίζω. Ευχαριστώ πολύ και τώρα τελευταίο ομιλητή είναι ο κύριος Γιάκοφτσίτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν αμφισβητώ τις καλές προθέσεις της Επιτροπής. Δεν αμφισβάλλω ότι έχετε καλές προθέσεις, κυρία Γιώροβα. Αυτό που προτείνετε συνιστά κάποια πρόοδο. Αλλά Δεν είμαι βέβαιος ότι επιτυγχάνατε το επιδεκόμενο αποτελέσματα. Και η ασπίδα προστασίας και το αλεξιβρόχιο είναι πολύ ωραίες συμφωνίες και πλέον έχουν και φάνταστα ονόματα. Το λέει και δεν είμαι σίγουρος ότι επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αποτέλεσμα όπως είπα, και νομίζω ότι ενδιαφέρονται οι Αμερικανοί πολίτες σε τελευταία ανάλυση κατά την πλειονότητά τους για τα δικά μου προσωπικά δεδομένα. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην προστασία των δεδομένων των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Πάντοτε είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε μεταξύ μας και για μένα προσωπικά για τους συναδέλφους αποτελεί έμπνευση η συζήτηση. Έχετε δίκιο ότι οι ροές δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις ΗΠΑ είναι πραγματικά τεράστια και πρέπει γρήγορα να φτιάξουμε ένα νέο σύστημα που θα προστατεύει τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών. Όχι λόγω των εταιριών που χρησιμοποιούν ε, αυτά τα στοιχεία ως βάση για τις δικές τους δραστηριότητες, αλλά επειδή όπως αναφέρθηκε ε, πρόκειται και για ε, καταστροφή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί παραμένουν σε νομική αβεβαιότητα. Είναι μια περίσταση κατά την οποία, έπρεπε να, την οποία μάλλον έπρεπε να λάβουμε υπόψη όταν έπρεπε να εργαστούμε για αυτό το θέμα μετά από την απόφαση του 10 αλλά και πριν. Χρειαζόμαστε βεβαίως εξασφαλίσεις και διαβεβαιώσεις από πλευράς των Αμερικανών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την νομική βεβαιότητα και να θέσουμε τέλος στις αβεβαιότητες γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σκέφτηκα την κατάστασή μας με τι σκέφτηκα ότι πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές οι διπλωματεύσεις μέσα σε εμπιστοσύνη και με δυνατότητες ελέγχους να πείσουμε τους Αμερικανούς μας ε, εταίρους ότι πρέπει να τηρήσουν την νομοθεσία τους και αυτά στα οποία ήδη δεσμεύτηκαν στις επίσημες επιστολές που υπογράφηκαν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Θα σας πω σήμερα ότι δεν μπορώ να πω ότι η ασπίδα προστασίας ως μηχανισμός για την προστασία των στοιχείων, της Ευρωπαϊκής, των, στοιχείων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απόλυτα τέλεια. Δεν μπορεί να είναι τέλεια και ούτε και εγώ θα είμαι απόλυτα ικανοποιημένη ποτέ. Γιατί υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα. Ένας από αυτούς είναι το θέμα της αμερικανικής νομικής τάξης που τόνισε πολύ σωστά ο κ. Άλμπρεχτ. Δεν έχουμε καμία εμείς αρμοδιότητα να αλλάξουμε την Αμερικανική νομοθεσία. Αλλά όπως σας είπα θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα αυτό της ΕΠΑ και έχουμε επανειλημμένα εκφράσει την πεποίθησή μας ότι τα στοιχεία θα προστατευτούν καλύτερα στην Αμερική εφόσον προστατεύονται εφόσον έχουν τη δικό τους δική τους νομοθεσία προς, περί προστασίας δεδομένων. Δεύτερος αντικειμενικός λόγος είναι η πρόσβαση στα δεδομένα για λόγους εθνικής ασφάλειας. Δείτε την κατάσταση στην Ευρώπη. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ζητήσει από τις μυστικές υπηρεσίες να είναι πιο διαφανείς και να ενημερώνουν τον κόσμο για το αν χρησιμοποιούν ή όχι αυτά τα στοιχεία. Ούτε καν ένα κράτος δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα. Θέλουμε κάτι, θέλαμε κάτι τέτοιο όταν διαπραγματευόμασταν με τη ΣΥΠΑ. Υπάρχουν όρια όμως. Πρέπει να σας το πω ανοιχτά. Δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι υπό την έννοια ότι έχουμε πετύχει το maximum που μπορούσαμε. Αυτό το οποίο όμως είναι πιο σημαντικό είναι ότι δεν θα πρέπει να μείνουμε επαναπαυμένοι για το μέλλον. Ε, ε, θα πρέπει να επαγρυπνούμε γιατί η Κομισιόν έχει δεσμευθεί, εγώ δεσμεύτηκα, οι συνάδελφοι δεσμεύτηκαν να παρακολουθούμε διαρκώ τι γίνεται στη ΣΥΠΑ και θα το κάνουμε αυτό με πολύ διαφανή τρόπο και στι ετήσιές μας εκθέσεις όπου αναμένουμε όλοι να συμβάλλουν με αξιόπιστα στοιχεία που θα δείχνουν την εξέλιξη της κατάστασης. Ε, και για την Αμερική και για την Ένωση. Αυτή η αναθεώρηση καθώς και η πολύ ισχυρή ρήτρα αναστολής είναι πολύ ε, στεναρή ασφαλιστική δικλίδα και δεν χρειάζεται sunset ε, clause όπως προτάστηκε. Ε, η κυρία Ιντεβέλτ είναι απόλυτα, έχει απόλυτο δίκιο. Η απόφαση ΣΡΕΜΣ μας καθοδήγησε, την περιμέναμε. γιατί ήμασταν πεπισμένοι ήδη πριν ε, βγει η απόφαση ότι η απόφαση αυτή θα μας έδινε τα επιχειρήματα αλλά και έναν πύχη με βάση τον οποίο να διαπραγματευτούμε μια σωστή ε, θέση, τη δική μας θέση. Και όντως έτσι συνέβη. Ε, ήμασταν ε, λοιπόν, ε, ακολουθήσαμε κατά γράμμα άρθρο προς άρθρο την απόφαση ΣΡΕΜΣ και διαπραγματευτήκαμε πολύ σκληρά με τους Αμερικανούς μας εταίρους, πάντοτε παραπέμποντας την απόφαση του δικαστηρίου. Δεν, μπορούμε, δεν μπορώ να είμαι βέβαια για το ότι αυτή η απόφαση, η επόμενη μάλλον, δεν θα είναι τόσο σοβαρή όσο η επόμενη, αλλά είμαι βεβαία ότι το σύστημα της ε, ασπίδας προστασίας θα μπορεί να προσαρμοστεί και στις επόμενες αποφάσεις του δικαστηρίου. Τώρα για τη Σύμφωνη Ομπρέλα. Δεν ε, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε κάτι μυστικό. Ένα σωρό γραπτές απαντήσεις στείλαμε στην Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ και θα θέλω, ήθελα να σας ζητήσω για να στηρίξετε όχι μόνο την ασπίδα προστασίας αλλά και την ε, Συμφωνία Ομπρέλα γιατί όπως είπα και πριν πρόκειται για βελτίωση της προστασίας των δεδομένων. Είναι αυτό και προς το συμφέρον των θυμάτων ποινικών ε, αδικημάτων ε, γιατί ενισχύουμε τους δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ένωση για θέματα ποινική δικαιοσύνης και ασφάλειας. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα θέματα ασφάλειας είναι ε, εξαιρετικά σημαντικά και ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να έχουμε καλύτερη, πιο ομαλή και πιο ασφαλή συνεργασία ανάμεσα στις αρχές τάξης της Ένωσης και τον ΗΠΑ. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να σας ζητήσω για τη στήριξή σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Um, thank you very much, Madam Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Και τώρα ε, ο Υπουργός κύριο έχει το λόγο. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Αποδεικνύεται ασφαλώς ότι δεν μπορούν να παραμείνουν ποτέ ανεξέλεγκτες οι ροές των δεδομένων και πάντα πρέπει να στηρίζονται και στην εμπιστοσύνη του πολίτη ότι τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται κατά τρόπο σύνομο τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στι ΗΠΑ. Εάν ο πολίτη έχει την ε, εντύπωση ότι δεν είναι σύνομη χρήση των δεδομένων του, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγείρει αντιρρήσει. Βέβαια βλέπουμε και από τη σημερινή συζήτηση πόσο μεγάλη σημασία έχει η απρόσκοπτη ροή δεδομένων και για τι μεγάλες, και για επιχειρήσεις και για την Αμερικανική διοίκηση αλλά και για, τους, ε, για την Ευρώπη. Θα μπορούμε δηλαδή να έχουμε πιο αποτελεσματική δράση, καταρχάς οι επιχειρήσεις ε, τόσο στην ε, Αμερικανική όσο και στην Ευρωπαϊκή πλευρά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Μπορούμε ταυτόχρονα να καταπολεμήσουμε το έγκλημα πιο αποτελεσματικά και να ενισχύσουμε την ασφάλεια και στις δύο υπήρους. Και πολλές ήταν οι ερωτήσεις που διατυπώθηκαν σε σχέση με την ε, προστασία των δεδομένων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι η ίδια η συμφωνία δεν συνιστά νομική βάση για την διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, μόνο συμπληρώνει άντλες συμφωνίας με μια διασφαλιστική δικλίδα για τα προσωπικά δεδομένα. Και αυτό έχει την σημασία του. Και βέβαια η συμφωνία μπορεί, εάν αποδειχθεί ότι δεν τηρείται ορθά από τα μέρη, να ε, πάψει να ισχύει, να ανασταλεί. Ε, ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό είναι αυτό ενός δικαστικού μηχανισμού που μπορεί να μην αποτελεί αυτή τη στιγμή γιατί δεν υπάρχει πραγματική νομική προστασία, δεν υπάρχει ένας πραγματικός δικαστικός μηχανισμός, αλλά υπάρχει ένας μηχανισμός του διαμεσολαβητή που πιστεύω ότι ειλικρινά θέλουν να δημιουργήσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε και να επιτρέψουν να λειτουργήσει κατά τον ορθό και προσήκοντα τρόπο. Βέβαια, ο διαμεσοπολιβαλληλαβητής δεν ζει σε κενό αέρος και δεν λειτουργεί σε κενό αέρος, αλλά συνεργάζεται με τις εσωτερικές αριθμιστικές αρχές των υπηρεσιών που θα καλούνται να δίνουν απαντήσεις ε, και εξηγήσεις. Άλλωστε και σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη-μέλη υπάρχουν ε, αντίστοιχα συστήματα επιτήρηση από ένα είδους ombudsman για τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων σχετικών με τις υπηρεσίες πληροφοριών ή χρήσιμες υπηρεσίες πληροφοριών. Ήταν μια σημαντική όμως συμφωνία, σε αυτό θέλω να καταλήξω. Μας εξασφαλίζει ένα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας βέβαια μόνο εάν τηρούνται οι προδιαγραφές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας από την τρίτη χώρα. Εάν η τρίτη χώρα προβαίνει σε μια αδιάκριτη και μαζική συλλογή δεδομένων, τότε δεν τηρούνται αυτές οι προδιαγραφές και αυτό έχει καταστεί απόλυτο σαφές στις επαφές μας με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ. Πρέπει λοιπόν και να λειτουργεί με βάση τους κανόνες και να έχει τα συστήματα επιτήρησης και εποπτείας το σύστημα αυτό, ώστε να μην γίνονται αδιάκριτες και μαζικές συλλογές δεδομένων. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνεται η διαλογή των δεδομένων λοιπόν και όχι μαζική τους ε, συλλογή και διακράτηση που μπορεί να γίνεται μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις και εφόσον ε, υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Επίσης για τη ρήτρα εκπνοή, τη ρήτρα sunset, ε, δεν θέλω να συμπληρώσετε τα περισσότερα στα όσα είπε η Επίτροπος. Είναι ζήτημα που απασχολείται τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το γνωρίζω. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Φως ότι δεν χρειάζεται εφόσον υπάρχει δυνατότητα της ε, ε κατέτος αναθεώρησης και εξέτασης του τρόπου λειτουργίας συμφωνίας δεν χρειάζεται ρήτρα εκπνοής. Επίσης ε, και η ασπίδα προστασίας αλλά και η συμφωνία του Αλεξιβροχίου μπορεί να προσφέρει επαρκή προστασία στους πολίτες μας και στα δεδομένα τους. Το καλύτερο, λέμε, πάντα είναι ο εχθρό του καλού. Βεβαίω είναι απαραίτητο να λειτουργήσει καλά το σύστημα αυτό, είναι απαραίτητο του πολίτε όπω και για τι επιχειρήσει. Και βεβαίω ελπίζουμε στην συνένεση του Κοινοβουλίου κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται έτσι